<clears throat> Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Θα σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα των εκλογών. Ήδη το αποτέλεσμα των εκλογών για το αξίωμα του Αντιπροέδρου. 703 ήταν η ψήφοι. Άκυρα 14. Αυτό σημαίνει πως τα έγκυρα ήταν 689. Η απόλυτη πλειοψηφία άρα είναι στα 300, στις 345 ψήφους. Θα σας δώσω τώρα τον αριθμό που έλαβαν οι υποψήφοι με αλφαβητική σειρά. Άλβαρο 199 ψήφισαν. Για την κυρία Αντζελίλη. 316. Ντιρόν. 182. Κάρας. 305. Μαρτίνες Μαρτίνες. 276. Μακμίλαν Σκοτ. 225. Κύριος Παπαστάμκος.

Βλάζακ 196 και Βίλαντ 268. Διεπιστώνω πως κανένας δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη απόλυτη πλειοψηφία. Γι' αυτό απαιτείται δεύτερος γύρος. Ερωτώ τους υποσφίους εάν όλες τους και όλοι τους είναι υποψήφοι για δεύτερο γύρο. Θα ρωτήσω ως εξής. Υπάρχει κάποιος ο οποίος αποσύρει την υποψηφιότητά του. Όχι. Οπότε θα έχουμε τον ίδιο κατάλογο υποψηφίων στο δεύτερο γύρο. Όλοι λοιπόν θα παραμείνουν και περνάμε στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας. Παρακαλώ τους ε, ψηφολέκτες να λάβουν τις θέσεις τους. Τυπώνονται τα ψηφοδέλτια. Τα αναμένουμε από στιγμή στιγμή. Παρακαλώ όμως ψηφολέκτες να πάνε στι θέσεις τους. Παρακαλώ λίγη υπομονή μέχρι να εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια. Με ειδοποιούν ότι εκτυπώθηκαν. θα ξαναρωτήσω. Είναι στη θέση τους οι ψηφολέκτες. Θα ξαναδιαβάσω τα ονόματα. Frau Borsellino, Herr Κύριε Βασουλίνο, κύριο Σόγκουρ, Παναγιώτοφ, Ποκ, κύριος Μπάγκο, ο κύριος Καλινόφσκι, ο κύριος Κάλβιν και ο κύριος Περέγιο Ροντρίκες. Παρακαλώ πηγαίνετε στις κάλπες. Αλλιώς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και σας παρακαλώ ειδοποιήστε με όταν φτάσετε στις κάλπες. Darf ich noch mal Οι ψηφολέκτες λοιπόν είναι στις θέσεις τους. Κάντε μου ένα νόημα. Μπορείτε να μου πείτε εάν οι ψηφολέκτες είναι στις θέσεις τους. Okay? It's okay? Yeah? Ναι. No. The member not. Frage nochmal. Θα ξαναρωτήσω. Είναι στις κάλπες, σε όλες τις κάλπες οι ψηφολέκτες. Ποιος λείπει. Frau Borsellino ist da. Herr Sogor. Κύριε Μπορσελίνο, Ζόγκουρ. Κύριε Ζόγκουρ. Herr Παναγιώτοφ. Κύριε Παναγιώτοφ. Ο Ποκ. Herr Μπάγκουπ. Κύριος Ο κύριος Κάλβιν. Κι όμω εκεί είναι. Παρακαλώ λοιπόν τώρα του κλητήρε να μοιράσουν τα ψηφοδέλτια. Παρακαλώ μοιράστε τα ψηφοδέλτια. Ich glaube, meine Damen und Herren, zur Prozedur brauche ich nichts mehr zu sagen. Δεν χρειάζεται να πω, πιστεύω, τίποτα άλλο για τη διαδικασία. Είναι η ίδια με τον πρώτο γύρο. Μπορείτε να σταυρώσετε 14 υποψηφίους. Παραπάνω σταυρή και είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο εάν δεν σταυρώσετε κανέναν επίσης. Die Abstimmung ist eröffnet. Άρχεται η ψηφοφορία. qui c'est le résultat sera publié ce soir. Απόψε δημοσιευθούν τα αποτελέσματα. Αλλά αν υπάρξει και τρίτος γύρος θα γίνει αύριο. Ja, ja. Dritte Wahlgang ist morgen. Ναι, ναι. Τυχόν τρίτος γύρος αύριο. Το αποτέλεσμα θα το μάθουμε απόψε.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 Darf ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer fragen, ob sie... Ψήφισαν οι ψηφολέκτες. Did the assessors vote? The assessors voted. Yeah, or they are on the road to vote. Ψήφισαν ή ψηφίζουν όπου να είναι. Ψήφισαν ο έδωσαν τα ψηφοδέλτια και ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Ja, bitte, Sie haben eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Παρακαλώ, έχει να πείτε κάτι από τη διαδικασία. Presidente, non propriamente un richiamo. Πρόεδρε, δεν επικαλούμε το κανονισμό, αλλά είναι πίστευτο μία περίοδος ε, στο Κοινοβούλιο όπου δεν εγγυέται η μυστικότητα της ε, ψήφου. Είναι αδιανόητο να ψηφίζει κανείς σε τόσο πολυπληθή αίθουσα με συναδέλφους που μπροστά πίσω δεξιά και αριστερά έχουν τη δυνατότητα να δουν αυτό που ο διπλανός ε, συνάδελφος ψηφίζει. Σε κάθε κοινοβούλιο τη στιγμή της ψηφοφορίας εκαθίστανται ε, καμπίνες, ε, ε κάποια διαχωριστικά που να μπορεί να ψηφίσει κανείς ξεχωριστά. Δεν το ζητάω να γίνει αύριο η ψηφορία αύριο, αλλά παρακαλώ στο μέλλον να ληφθεί υπόψη αυτή η παρατήρησή μου. Να μπορώ να το πω το παραπάνω. Μάλιστα, το σημειώνω. Ξαναρωτάω, κυρίε και κύριοι, ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν και οι ψηφολέκτε. Εντάξει,